καμία αντίρρηση και άρα διακόπτεται η Σύνοδος Ολομελίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Σας εύχομαι καλό ταξίδι. Λύεται η συνεδρίαση. thank you.